Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε την απογευματινή συζήτηση, ε, καλωσορίζω τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ. Τον συγχαίρω επίσης για τα θαυμάσια αποτελέσματα που πέτυχε στο Βουκουρέστι την περασμένη εβδομάδα. για το, την Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Συγχαρητήρια και ας ξεκινήσουμε. Περνώντας τα πολωνικά, τη γλώσσα μου, ξαναρχίζουμε τη συζήτηση και το πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση για τις αγορές στα χρηματοπιστωτικά μέσα ε, η έκθεση του κυρίου Φέρμπερ και η άλλη έκθεση του κυρίου Φέρμπερ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποίηση του κανονισμού ΕΜΗ σχετικά με τα εξοχρηματιστηριακά παράγοντα, τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μάρκους Φέρμπερ. Είμαι εισηγητή και για τι δύο εκθέσει. Τέσσερα λεφτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Νομίζω ότι με τη σημερινή συζήτηση για το MIFID έχουμε μπει στην ουσία ε, των ρυθμίσεων των χρηματαγορών και των χρηματοπιστωτικών μέσων γιατί αυτό θέλουμε, να ρυθμίσουμε τις χρηματαγορές ολόκληρες, όχι με μονομένα προϊόντα όπως κάναμε στο παρελθόν. Ε, μερικά κλειδιά μόνο θα σας αναφέρω. Πέρυσι δυσκολέψαμε τη ζωή μας. Στην Επιτροπή μας κάναμε ακρόαση ολόκληρη ε, όλους τους ενδιαφερομένους, ρωτήσαμε όλες τις ε, ομάδες ε, ενεχομένων και στη συνέχεια με διάφορα έγγραφα εργασίας, διαδικασίες και τα λοιπά καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα που έρχεται ε, και στη συζήτηση σήμερα και αύριο στην ψηφοφορία. Θέμα υπαριθμών 1. Η δομή και η διάρθρωση της αγοράς. Οπότε θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια στις χρηματαγορές έχουν αλλάξει πράγματα και είναι προς το συμφέρον μας και του Κοινοβουλίου ε, να ε, γίνεται οποιαδήποτε συναλλαγή εντός των πλαισίων MIFID. Γι' αυτό υπάρχουν όλες αυτές οι ε, ε διατάξεις για τους μηχανισμούς ε, οργανωμένης διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένες διατάξεις, με συγκεκριμένες συναλλαγές και διάδραση των πελατών μεταξύ τους. Θα πρέπει λοιπόν έτσι και πιστεύω ε, να συνεισφέρουμε ε, έτσι ώστε όλα αυτά τα έγγραφα, τα έξω χρηματιστριακά παράγωγα να είναι αντικείμενο συναλλαγής εντός του MIFID. Κάτι άλλο που δεν είχαμε λάβει υπόψη μας ήταν οι λεγόμενες αλγοριθμικές συναλλαγές και εδώ χρειάζονται σαφείς κανόνες του παιχνιδιού γιατί ε, αυτός ο τομέας μπορεί να είναι άκρος επικίνδυνος και πολλές φορές υφίσταται και χειραγώγηση και αυτό θα πρέπει λοιπόν να υπόκειται σε καθεστώς με προθεσμίες, με δυνατότητες ε, διακοπής της συναλλαγής, με δυνατότητα δοκιμής και εποπτείας και οι εποπτικές δομές να κοιτάνε τους αλγορίθμους και να υπάρχουν ε, και ελάχιστες τιμές και ειδικά καθεστώτα και ειδικά τέλη που θα πληρώνουν οι συναλλασσόμενοι. Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι οι προθεσμιακές συναλλαγές. Ε, ε, ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη κερδοσκοπία και θέλουμε να τα περιορίσουμε αυτά για να μην κάνουμε λάθος ρυθμίσεις και να μην μπορεί ε, κάποιος στον τρίτο και στον τέταρτο κόσμο να αγοράζει εμπορεύματα. Εδώ πρόκειται λοιπόν για τις αγορές εμπορευμάτων ε, χωρίς να υπάρχει ε, πρόβλημα στην πραγματική αγορά με ανώτατες τιμές ε, για ε, τέτοια δικαιώματα, αλλά κάποιος που μπορεί να αποδείξει ότι χρειάζεται ένα ε, εμπόρευμα με το λεγόμενο έλεγχο της ε, θέσης, ε, position check, να μπορεί να γίνεται. Και η προστασία των επενδυτών μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επιλέξαμε μια πολύ μεγάλη ευρύτατη προσέγγιση για την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών. Υπάρχουν ομάδες πελατών που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Ο κάθε μικροεπενδυτής και μικροκαταθέτης δεν πρέπει αναγκαστικά να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα πολύ περίεργα και περίπλοκα δομημένα προϊόντα. Επίσης ε, να γίνονται έλεγχοι και με τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και ε, με υποχρέωση δημοσίευσης, αλλά ε, είναι και θέμα επικουρικότητας. Τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις δομές τους και τα συστήματά τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αντίστοιχες προσαρμογές. Και εκεί νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Επειδή τέλειωσε και ο χρόνος μου, να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνεισέφεραν στην ε, προσπάθεια. Ε, κρίμα που για ένα τόσο δύσκολο θέμα έχω μόνο τέσσερα λεπτά ω εισηγητή. Ευχαριστώ όλου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επικοδομητικό τη ρόλο του τελευταίου μήνε και εβδομάδε και ελπίζω αύριο να βγει ένα ισχυρό αποτέλεσμα από την ψηφοφορία και να μπορέσουμε να πάμε σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ε, το συντομότερο όσο γίνεται να κλείσει αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιο συγκεκριμένα στον Επίτροπο Μπαγνιέ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η σημασία της εβδομάδας της εσωτερικής αγοράς είναι πολύ σημαντική και για τα κεφάλαια. Ε, την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια ενδελεχή συζήτηση. Τώρα μιλάμε για ένα μείζον θέμα που είναι ακρογωνίως λήθος. Ο Μάρκους Φέρμπερ το υπενθύμησε ε, στην ατζέντα για τις ρυθμίσεις. Ε, συχνά δείχνω αυτό τον πίνακα στου Υπουργού και στου αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τα 29 κείμενα που κινητοποιούν την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚΟΝ με την πρόεδρο κυρία Μπόλς, τους ε, συντονιστές της, ε, τον εισηγητή και του κοιόδη εισηγητέ. Αυτός ο λίθο ε, είναι για την ενία για τις χρηματαγορές, είναι ότι κάνουμε για την ενιαία αγορά Κάνουμε επίσης προσπάθειες και για τον τραπεζικό τομέα, ούτως ώστε σε όλο το χρηματοπιστωτικό τομέα να έχουμε την απαραίτητη διαφάνεια, την ευθύνη, την ασφάλεια για τους επενδυτές και τους αποταμιευτές. Χωρίς να αφήσουμε καμία θέση στην ρυθμιστική διαμεσολάβηση, στο αρμπιτράζ, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς απέναντι στους άλλους εταίρους του G20. Ε, σας ευχαριστώ για αυτή την προσπάθειά σας κύριε Φέρμπερ. Ε, που όπως είπατε ο στόχος μας είναι να ξεκινήσει πολύ γρήγορα η συζήτηση του τριμερούς διαλόγου. Για το ΜΕΦΙΝΤ έχουμε τους ίδιους ε, στόχους. Η έκθεση που ετοιμάσατε, κύριε Φέρμπερ, ενισχύει και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, για τη ε, διάρθρωση για τη δομή της αγοράς. Και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουμε σαν στόχο οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης, είτε πολυμερής είτε διμερής, να γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον ε, διαφανές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έβαλε έναν ορισμό της αγοράς μαζί με μια υποχρέωση διαπραγμάτευσης για τις ε, πλατφόρμες εκτέλεσης που είναι διαφανείς για τις συναλλαγές μικρού, μικρής κλίμακας, πούμε, τις μικρές συναλλαγές. μπορούμε επίσης να καταργήσουμε την κατηγορία του OTF για την αγορά των μετοχών. Αυτό θα πρέπει όμως να το αναλύσουμε με μεγάλη προσοχή. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις συνέπειες μια τέτοια τροποποίηση σε σχέση με τη δική μας πρόταση. Αν περιορίσουμε την πολυμερή διαπραγμάτευση μόνο στην ρυθμιζόμενη αγορά και στις πλατφόρμες MTF, τις τον πολυμερή δηλαδή μηχανισμό διαπραγματεύση, δεν μεταρρυθμίζουμε την κατάσταση όπω έχει σήμερα, που επιτρέπει ας πούμε στου τρέιντερ υψηλή συχνότητα σήμερα να διασταυρώνουν τους εντολέ του με αυτέ των επενδυτών. Χωρί αυτό βέβαια, να να χωρίς οι επενδυτέ να μπορούν να πούν τίποτα. Χωρίς, ε, πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε να περιορίσουμε τόσο πολύ το πεδίο εφαρμογή των οργανισμένων α, μηχανισμών διαπραγμάτευσης. Επίση, για τι συναλλαγέ ε, υψηλή συχνότητα. αν θέλουμε οι συναλλαγές να πάνε σε πλατφόρμες ε, διαπραγμάτευσης πολυμερής και διαφανής, θα πρέπει καλύτερα να πλαισιώσουμε την ε, διαπραγμάτευση ψηλής συχνότητας που την προτιμούν σε αυτές τις πλατφόρμες. Εδώ λοιπόν συμφωνούμε και συμμεριζόμαστε τους ίδιους στόχους. Το κείμενο είναι η ευκαιρία για να ξαναδούμε τους κανόνες για το high frequency trading, για την διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας. Είμαι έτοιμος να αναγνωρίσω μια κάποια χρησιμότητα ε, στη διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας για να εξασφαλίσει ρευστότητα. Αλλά αναμφίβολα, θα, παράλληλα, υπάρχει και ένας εγγενής ε, κίνδυνος για τις αγορές εξαιτία της. Στον τραπεζικό τομέα κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια για να εποπτεύσουμε και να μειώσουμε αυτού του είδους τον κίνδυνο. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι στον τομέα των αγορών. Ακριβώς γι' αυτό η Κομισιόν πρότεινε ένα σύνολο πολύ συγκεκριμένων κανόνων για να πλαισιώσει, πλαισιώσει και να υπευθυνοποιήσει αυτούς τους φορείς και παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν και έγκριση και να υποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές και θα πρέπει επίσης να δεσμεύονται να δίνουν την απαραίτητη ρευστότητα στις αγορές. Ευχαριστώ πραγματικά τον εισηγητή τον κύριο Φέρμπερ που πρότεινε να διατηρηθούν αυτά τα σημεία και υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να προωθεί αυτή τη συζήτηση και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε διεθνή φόρουμ, ούτω ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ίσων ευκαιριών, ίσων κανόνων. Ε, τρίτο σημείο, ε, η αγορά των παραγόγων στα βασικά εμπορεύματα. Είναι διαφορετικές αυτές οι αγορές, γιατί καλή τους λειτουργία σημαίνει επηρεάζει την καθημερινότητα όλων των καταναλωτών. Και ξέρουμε ότι σε ορισμένε αναπτυσσόμενε χώρε αφορά και την επισητιστική ασφάλεια ενός ε, μεγάλου τμήματος του πληθυσμού τους. Ε, η κερδοσκοπία στις πρώτες και οι συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η κερδοσκοπία στην ε, επιστηστική ασφάλεια των χωρών αυτών είναι απαράδεκτη. Θέλω να υποστηρίξω ξεκάθαρα τις προτάσεις σας που σκοπό έχουν να ενισχύσουν το καθεστώς για τον περιορισμό της θέσης, διατηρώντας τη δυνατότητα για τις εμπορικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτές τις αγορές όταν πρόκειται για θέματα εγγύησης, κάλυψης. Τέταρτο σημείο, εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος για την παραρχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Και εδώ είμαι ικανοποιημένο που η θέση μα την χάνει υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι αυτό το καθεστώ είναι το καλύτερο για να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική ρύθμιση των αγορών και να περιορίσει τον κίνδυνο ε, ρυθμιζόμενης διαμεσολάβησης, αρμπιτράζ. Ε, επίσης ε, το συζητάμε και στο G20 και στο Financial Stability Board. Αυτή η σημαντική συζήτηση ε, μου δίνει ευκαιρία να αναφέρω δύο-τρία θέματα διαφορετικά, τηλεγραφικά όμως, που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, γιατί θα πρέπει να έχουμε πολύ σημαντικές απαιτήσεις κανονιστικές και ρυθμιστικές. Καταρχάς, η προσυναλλακτική διαφάνεια, θα πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί, να μην πάρουμε το ρίσκο ε, με συγκεκριμένες διατάξεις, να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιου φορείς να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται μέσα σε ένα νέφος ε, χωρίς καμία διαφάνεια. Θα πρέπει να είναι το ίδιο επίπεδο διαφάνειας, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο καθένας και ανεξάρτητα από το είδος του επενδυτή, από το, το εύρος, την ευρωστία του κτλ. Αν είναι ιδιώτης ε, Η προστασία των επενδυτών, άλλο θέμα. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μια νομοθεσία που βελτιώνει τις συνθήκες επενδύσεων, ε, διευκρινίζοντας τους ρόλους και τα οικονομικά συμφέροντα κάθε μέρους. Ακριβώς για αυτό το λόγο τον επανέλθουμε σε μια απλή πληροφόρηση σε της Επιτροπής των Ενδιαμέσων δεν νομίζω ότι εγγυάται την προστασία των επενδυτών ούτε ε, μας εξασφαλίζει το επαρκές επίπεδο ανεξαρτησίας. Η πρόταση που κάναμε ε, να σταματήσουμε ε, την ίσπραξη τελών για τις ανεξάρτητες συμβουλές εξασφαλίζουν μεγαλύτερη και ανεξαρτησία και διαφάνεια και είναι ο μόνος τρόπος για να προσελκύσουμε υγιείς επενδυτές και υγιείς επενδύσεις. Θα πρέπει επίσης να διατηρήσουμε τις απαιτήσει μας σε ό,τι αφορά τη δέσμη των μέσων που θεωρούνται μη περίπλοκα. Ε, το να το διευρύνουμε πολύ σημαίνει ότι βάζουμε και προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα και πολλούνται αναγκαστικά στους ε, επενδυτές. Τρίτο σημείο, τελευταίο σημείο μάλλον, ε, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις. Για να έχουμε υγιή ανταγωνισμό ε, στην μετασυναλλακτική αγορά είναι απαραίτητο για να έχουμε μια πραγματική ενιαία αγορά και να εμποδίσουμε υπερβολικά ψηλή ε, συσσόρευση κινδύνων σε μονοπωλιακές αγορές. Αυτά κύριοι και κυρίες βουλευτές. Ε, ο διάλογος συνεχίζεται μεταξύ μας. Άκουσα τα λόγια του, του κυρίου Φέρμπερ. Είμαι στη διάθεσή σας κύριε Φέρμπερ και εγώ και η ομάδα μου, οι συνεργάτες μου, ούτως ώστε να καταλήξουμε με ένα φιλόδοξο σχέδιο, γιατί η νομοθεσία αυτή είναι πολύ σημαντική νομοθεσία για το MIFID. Θα πρέπει μαζί να βρούμε μια καλή ισορροπία, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, εμπιστοσύνη των επενδυτών. Και έχω εμπιστοσύνη στην κοινή μα δράση για να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Εκ μέρου τη Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνα και ενέργεια. Ο κύριος Κράμερ. Ο δικός μου ρόλος σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση της ρύθμισης ε, των χρηματαγορών περιορίζεται στα θέματα βιομηχανίας, γιατί εξ ονόματος η Επιτροπής Ήτρε μιλώ. Γιατί ε, βεβαίως χρειάζεται να ρυθμιστεί η χρηματαγορά, αλλά υπάρχει και μεγάλος ακτιβισμός εδώ, ε, σε αυτή τη ρύθμιση. Και για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κανονικά με θέματα ε, ορισμών και ερμηνεών μπορεί η πραγματική βιομηχανία να ε, θυγεί. Ας πούμε, ε, ε, όταν έχουμε μικρές επιχειρήσεις, αστικές, ε, δημοτικές εταιρείες στη Γερμανία ή μικρούς γεωργικούς συνεταιρισμούς, δεν θα πρέπει να θεωρούνται τράπεζες και να έχουν υποχρεώσεις ας πούμε παράδοσης με συγκεκριμένες αυστηρές ημερομηνίες. Αυτό θα ήταν μια παράπλευρη απώλεια της παρούσης ρύθμισης που δεν θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον κανενός. Κατά την άποψή μου οι ε, βιομηχανικές εταιρείες θα πρέπει να έχουν άλλη αντιμετώπιση από ότι τραπεζικές εταιρείες ε, κάνουν ε, συμβόλαια ανταλλαγής εμπορευμάτων όχι για λόγους κερδοσκοπίας αλλά για λόγους πραγματικής εξασφάλισης. Δεν γνωρίζω καμιά εταιρεία ούτε παροχής ενέργειας ούτε εμπορική που να τηρεί αυστηρά όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφής. Τελικά καταφέραμε να λάβουμε υπόψη μας το τελικό νομοθετικό πακέτο και αυτές τις πτυχές και νομίζω ότι αυτό το δευτερεύον που μπορεί να είναι δευτερεύον για τη χρηματαγορά αλλά είναι σημαντικό για τη βιομηχανία ρυθμίστηκε σωστά. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και τώρα ερχόμαστε στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Στόλογιαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φέρμπερ για τις ε, δύο εκθέσεις του. Όλα τα μέλη της Επιτροπής, Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής υποστήριξαν τις δύο αυτές εκθέσεις και περιμένουμε και ελπίζουμε ότι και η Ολομέλεια θα τις υπερψηφίσει με ευρία πλειοψηφία. Τα συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα ε, κλείνουν ορισμένα παραθυράκια της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην χώρα μου, τη Ρουμανία, ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο με συναλλαγές ε, χρηματοπιστωτικών μέσων σε αδιαφανή αγορά και μη ρυθμιζόμενη αγορά. Ε, οι επενδυτές ε, έχασαν πολλά χρήματα και η ρυθμιστική αρχή έχασε ε, πολύ από το κύρος του, της. Οι επενδυτές δεν είναι εύκολο να καταφύγουν στα δικαστήρια, να προσφύγουν σε δικαστήρια σε τέτοιου είδου περιπτώσει. Και γι' αυτό το λόγο θα υπερψηφίσω τις δύο αυτές εκθέσεις. Θεωρώ ότι οι εξωχρηματιστηριακές αγορές, καθώς επίσης και άλλες πλατφόρμες και μηχανισμοί συναλλαγών θα πρέπει να γίνουν πιο διαφανείς. Ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περισσότερο τα συμφέροντα των επενδυτών. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Μάρτιν για σας. Δέχεστε κύριε Στολογιάννη. This is behind you. Okay, so please, Mr. Martin, the floor is... Πίσω σας. Κύριε Μάρτιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Με ενδιαφέρον άκουσα τα όσα είπατε και σας παρακολούθησα. Έχω μια ερώτηση όμως. Για ποιο λόγο η δική σας πολιτική ομάδα, παρόλο που και ο εισηγητής δικό σας είναι, και τα είπε αλλιώς, γιατί συμφώνησε με αυτό το συμβιβασμό για τις προβλέψεις, ε, αντί να βεβαιωθείτε ότι το κόστος δεν θα μετακυληθεί στον τελικό ε, καταναλωτή για τις προμήθειες. Ναι, πώς ε, τα καταφέρατε έτσι τελικά και βγήκε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμούσατε. Thank you. I'm not so clear that... Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή. Με χαρά μου θα την υποστήριξω το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές ο κύριος Γκέμπελς. Κύριε Πρόεδρε, έχω 120 δευτερόλεπτα για να εκφράσω την συνένεση της ομάδας μου για τη συμφωνία. Ε, η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβαση ε, από τι ευρωπαϊκέ ρυθμιστικέ αρχέ και τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ για να αποφύγουμε οποιαδήποτε καταχρηστική και καταστρεπτική κερδοσκοπία. Τα συμφέροντα των καταναλωτών προστατεύονται περισσότερο. Ε, η διαφάνεια είναι λέξη κλειδί. Διαφάνεια για τις τιμές χάρη στην επικουρικότητα, τα κράτη-μέλη δίνουν επιπλέον περισσότερες επιλογές μέχρι και την απαγόρευση των αντιπαροχών. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη και να προτείνει και διορθώσεις. Επίσης, οι προτάσεις σας βάζουν φραγμούς ε, στην κερδοσκοπία των αγορών βασικών προϊόντων και των ε, γεωργικών προϊόντων. Οι φορείς αυτής της αγοράς θα είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ε, στοιχεία και υπάρχουν όρια για τις θέσεις που ένας φορέας ή μια ομάδα φορέων, ένας όμιλος μπορεί να έχει. Ένα βασικό στοιχείο είναι η πλαισίωση του, της διαπραγμάτευσης υψηλής συχνότητας και ε, η πληροφόρηση για τις τιμές της αγοράς. Όταν ε, μπαίνουν εκεί πέρα ε, οι υπολογιστές που εκτελούν εντολές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου ή δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου. Αυτή η διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας δεν δίνει καμία ρευστότητα στην αγορά για μερικά ε, δευτερόλεπτα, ούτε καν δευτερόλεπτα υπάρχουν αυτές οι εντολές. Μέχρι το 80%, το 80 ε, των εντολών ε, έχουμε α, σε μη α, υψηλή συχνότητα διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι εντελώς άπιαστες. το βασικό είναι να πλήξουμε του κερδοσκόπους και να προωθήσουμε του υγιεί επενδυτέ. Χρειαζόμαστε τις χρηματαγορές και θα πρέπει να εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Από τους φιλελεύθερους, ο κύριος Όλε Σμιτ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ τον Μάρκους Φέρμπερ για την πολύ επικοδομητική του δουλειά. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο, πάρα πολύ τεχνικό ε, και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ισορροπημένο συμβιβασμό. Έτσι βάζουμε τις βάσεις για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις χρηματαγορές και των καταναλωτών. Έχουμε βάλει κανόνες για την διαπραγμάτευση ψηλή συχνότητας, μειώντας το κίνδυνο που επισύρει, καθώς και την ανεξέλεγκτη λειτουργία των μηχανισμών διαπραγμάτευσης. Επίσης, ε, είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη κανόνων για τις ε, εθνικές αγορές, όπως της ε, Σουηδίας. Όπως είπε ο εισηγητής, το να υπάρχει επιλογή, το να υπάρχει καλύτερο ανταγωνισμός, το να υπάρχει πιο στεναρή αγορά κεφαλαίων, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Σε ό,τι αφορά τις αντιπαροχέ, τις προμήθειες δηλαδή που εισπράττονται. Νομίζω ότι η οδηγία δεν ήταν επαρκή για να αποτρέψει τις επιθετικές ε, συμπεριφορές. Εγώ ως φιλελεύθερο, θεωρώ ότι εδώ υπάρχει, κύριε Γκέμπλς, ένα πρόβλημα. Αυτή η γενικευμένη απαγόρευση των αντιπαροχών δεν νομίζω ότι είναι σωστή. Κατά την άποψή μας, κατά την άποψη των φιλελεύθερων, θα θέλαμε χώρε, όπως η Μεγάλη Βρετανία που θέλουν κανόνε πιο αυστηρούς να τους έχουν. Μία γενική όμως απαγόρευση σε όλη την Ευρώπη θα έχει ως αποτέλεσμα ότι όποιος έχει ένα χαμηλότερο εισόδημα δεν μπορεί να έχει πλέον ε, δωρεάν συμβουλές για τις επενδύσεις του. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν κάποιοι να αποκλειστούν από την αγορά. Η προσφορά χάρη στον ανταγωνισμό θα ενισχυθεί επίσης. Επομένω, οι συμβουλέ θα δίδονται σε όλου του καταναλωτέ. Αυτό είναι σημαντικό για να προστατεύσουμε καλύτερα του απλού αποταμιευτέ. Ευχαριστώ κύριε Φέρμπερ και ευχαριστώ όλου τους κοιόδης ηγητέ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ο κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία γενικά για την έκθεση αυτή σε κομβικά σημεία έχουμε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έφερε μεγάλα βήματα προς τη ε, σωστή κατεύθυνση και το βελτιώσαμε. Θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια στις δομές τώρα της αγοράς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αγορά παραγόγων, ε, στα πλαίσια της MIFID, οι αποφάσεις ε, για τις αλγοριθμικές συναλλαγές και ο συμβιβασμός μας είναι πολύ πιο προωθημένες από τις αρχικές Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής και αξίζουν την υποστήριξη και του Κοινοβουλίου γενικά. Και σε αυτά τα θέματα που γνώρισαν μεγάλη δημόσια κριτική έχει βελτιωθεί η έκθεση και σε ό,τι αφορά την κερδοσκοπία ε, στα εμπορεύματα και τα τρόφιμα, μετά πολύ δύσκολες συζητήσεις, ε, ενισχύσαμε το κείμενο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα όρια των θέσεων τώρα είναι πλέον δεσμευτικά και βεβαίως χρειάζονται και άλλες αλλαγές για να καλύψουμε και άλλα κενά που έχουν απομείνει και ελπίζω να συμπληρωθεί αυτό από την ψηφοφορία και τελικά από τον τριμερή διάλογο. Και χαίρομαι που ο κύριος Μπαρνιέ ήδη υποστηρίζει και δηλώνει ότι ε, ε, υποστηρίζει την θέση του Κοινοβουλίου. Εκεί που χωλαίνει η έκθεση είναι η προστασία των καταναλωτών. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα με να απαγορεύουμε κάποια προϊόντα και αυτό είναι πρόοδος, αλλά δεν έχει ε, μία πρόοδος γίνει για τις αντιπαροχές και την παροχή συμβουλό γιατί δεν προσανατολίζεται στον πελάτη η συμβουλή, αλλά στο ποιο προϊόν θα σου φέρει το μεγαλύτερο κέρδος και τη μεγαλύτερη προμήθεια στον πολιτή. Κοιτάξτε τι έγινε με τα ανοιχτά ταμεία ε, τα επενδυτικά και τα στεγαστικά. Ε, για τους πολίτες στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία ε, δεν αλλάζουν πολλά. Τα κίνητρα του πολιτή είναι κυρίως η προμήθεια και όχι η προστασία του καταναλωτή και θα ήθελα πιο ισχυρές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές η κυρία Σουίμπορν. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους συναδέλφους για τη δουλειά τους. Ένα από τα πιο, ένα από σημαντικά σημεία είναι η όρια για την διαφάνεια σε ε, μη μετοχικές αγορές. Ε, χαίρομαι που όλες οι ομάδες του Κοινοβουλίου υποστηρίζουν ένα κείμενο που ε, διευκολύνει ε, τις επενδύσεις σε αγορές ε, μετοχών εταιριών θα πρέπει οι εταιρείε να μπορούν να συλλέξουν χρήματα από αλλού εκτό των χρηματιστηρίων. Ε, η αγορά όμως, η διοδομή της αγοράς θα πρέπει ε, να προσαρμοστεί με καινούριου κανόνες διαφάνειας. Νομίζω ότι το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το κάνει αυτό. Και πιστεύω το ίδιο θα πρέπει να κάνει και το Συμβούλιο. Με απογοήτευσε όμω το ότι δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία για να εγγυηθούμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των επενδυτών για όλους τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη μας θα πρέπει να μπορούν να, ε, μπορούν να απαγορεύσουν όλες, κάποιο είδου προμήθεια. Είναι απογοητευτικό. Νομίζω, μπορείτε να να διαβάζετε λίγο πιο αργά διότι δεν μπορούν να σα παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Ε, το δικό μου κράτος και οι κατοχώρες έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζουν μια πλήρη απαγόρευση. Ελπίζω ότι και άλλα κράτη-μέλη θα το κάνουν. Ε, μια παρανόηση κοινή είναι ότι η μυφήντα φορά τις ε, διαπραγματεύσεις υψηλής συχνότητας. ε, αυτά έχουμε πολλές φορές συζητήσει την προστασία του καταναλωτή. Έχουμε περιλάβει ε, ε, μέτρα όπως ε, έλεγχο, εποπτεία των αλγορίθμων κλπ. με τρόπο που να μην εμποδίζει την ανάπτυξη τεχνολογίας. Αυτό θα δίνει και στους ιδιώτες και στους μακροπρόθεσμους επενδυτές την σιγουριά ότι δεν θα υφίστανται παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές. Επίσης όλα τα επιχειρηματικά ρολόγια θα πρέπει να δείχνουν την ίδια ώρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερο σύστημα εποπτείας. Με αυτόν τον τρόπο θα δουλεύουν όλοι μαζί στον ίδιο ρυθμό. Νομίζω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον για του επενδυτέ, μικρού και μεγάλου, και για τι εταιρείε που χρειάζονται ε, να δανειστούν χρήματα από τι αγορέ. από την ΚΟΕ, ο Γιώργαν Κλούτε. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία και ιδιαίτερα τον Μάρκους Φέρμπερ, τον εισηγητή. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία, ειλικρινής και σωστή. Δεν είναι δεδομένο αυτό στο Κοινοβούλιο και πραγματικά το εκτιμώ πολύ. Θα ήθελα όμως εδώ να ευχαριστήσω και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κερδοσκοπία ε, γύρω από τα τρόφιμα. Ε, ασχολήθηκαν πάρα πολύ και ο εισηγητή και θέλω να ε, το υπογραμμίσω, το δέχτηκε. Ούτε αυτό είναι αυτονόητο στο Κοινοβούλιο, ούτε εύκολε ήταν οι συζητήσεις, ούτε απλές και άνετες πάντα. Είναι σημαντικό όμως που ακούσατε και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις εδώ, γιατί το θέμα είναι αρκετά στριφνό και στεγνό, ε, τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο και οι πολίτες. Είναι σημαντικό και κάνει καλό και στο Κοινοβούλιο ένα τόσο σημαντικό θέμα να ε, έχει συμμετοχή και το Κοινοβούλιο σε αυτό. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Σβέν Γκίγκολτ. Ε, είναι καλό και σωστό αυτό που κάναμε για τη γερδοσκοπία στα τρόφιμα, αλλά παραμένουν ορισμένα κενά που θα πρέπει να καλυφθούν και ορισμένα παραθυράκια. Αυτό θα το δείξει η πείρα το πώς θα λειτουργήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αλγοριθμικές συναλλαγές, το υποστηρίζω και μπορώ να το ψηφίσω απολύτως ε, με όλη μου την καρδιά και η πολιτική μου ομάδα σε μεγάλο βαθμό. Ούτε αυτό είναι αυτονόητο. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι καλά τα πήγαμε για τις προμήθειες ε, και τις αντιπαροχές. Συμφωνώ, εδώ χρειάζεται λίγο κάποια βελτίωση και προσαρμογή, αλλά δεν είναι καθόλου απλή αυτή η ιστορία. Αύριο ε, υπάρχουν και κάποιες σχετικές τροπολογίες να δούμε τι θα βγει από την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από την Ελευθερία και Δημοκρατία ο κύριος Χέλμερ. Uh, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, εξασφαλίζει το 36% ε, των ε, χρηματαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε οι πρωτοπόροι στις χρηματαγορές και έχουμε κεντρικό ρόλο σε διάφορες συναλλαγές. Με τέτοιες λεπτομερείς ρυθμίσεις θα μας πλήττεται γιατί κάνετε τα εξοχρηματιστριακά προϊόντα λιγότερο ελκυστικά. Οι ρυθμιστικέ αρχές της Ευρώπης που ξέρουν αυτά τα θέματα το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Το να ξαναγίνεται όλες οι συναλλαγές να περνάνε μέσα από τα ε, χρηματιστήρια νομίζω ότι είναι προς το βλάπτη όλους τους φορείς. Το βασικό είναι να κλείσουμε τα παραθυράκια. Οι διαπραγματευτές ε, βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου με τις ρυθμιστικές αρχές. Ε, υπάρχει μία κίνηση προς τα κάτω, ενώ παράλληλα το εμπόριο ακολουθεί την δική του πορεία, ε, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία. Αυτή η προσέγγιση για φοβερές και λεπτομερείς ρυθμίσεις οδηγεί στην ύφεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς αυτές οι δύο εκθέσεις είναι ακόμα ένα καρφί στο, στο φέρετρο ε, των χρηματαγορών του Λονδίνου. Ε, Βερολίνο, ε, Βρυξέλλες, Φραγκφούρτη κτλ. Μας μισούν όλοι γιατί έχουμε επιτυχίες. Ευχαριστώ. Ωραία, για τις μία γραμμένες ο κύριος Μάρτιν. Ρότζερ, Ρότζερ, Ρότζερ. Και το εννοώ. Τι ήταν αυτό, δεν ήταν το τάδε έφη Ζαρατούστρα, ήταν τάδε έφη City του Λονδίνου. Το αντίθετο είναι το σημαντικό και το σωστό. Μίφιτ 1, Μίφιτ 2 είναι αφηρημένε έννοιε. Μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Δεν θυμάστε με ποια μορφή ο Επίτροπο κ. Μακρύβη ήρθε εδώ και ε, επιτέθηκε ε, στο Λονδίνο και τις άλλες χρηματαβορές και είπε τι θα κάνει η Μύφιτ 1. Και ο κύριος Μπαρνιέ λέει όχι έτσι, γιατί στο μεταξύ τι έγινε. Δύο τρεις, τρία, τρεις χάθηκαν στις δυνατότητες που υπήρχαν λόγω της υπορρύθμισης. Βεβαίως είναι μεγάλη πρόοδος η MIFID 2, δεν χωρά καμιά αμφιβολία, παραμένουν τα κενά. Ε, ακούστηκε γιατί έξω χρηματιστηριακά ε, παράγωγα υπάρχουν πολλές δυνατότητες ακόμα. Ε, και σε κάποιες άλλους ε, τόπους διαπραγμάτευση να φύγουν. Ε, σε αντίθεση με τα όσα είπε η G20 θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες όλα να ελέγχονται. Ο, ε, κάθε επενδυτής και εγώ δεν έχω καταλάβει σωστά οι δημοκράτες γιατί ψήφισαν τελικά αυτό για τις προμήθειε. Ποια συμφέροντα κρύβονται από πίσω. Οι πράσινοι ωραία τα είπαν. Το βασικό πρόβλημα είναι το σύστημα των αντιπαροχών και των κινήτρων. Δηλαδή, εάν οι ε, λάθος δραστηριότητες στην πραγματική οικονομία ανταμείβονται, καταλήγουμε εκεί που είμαστε. Στις αλγοριθμικές συναλλαγές είναι ε, σωστά αυτά που κάνουμε, αλλά παραμένουν πάρα πολύ λίγα. Ευχαριστώ. Επόμενοι ομιλητές. Δύο λεφτά. Ε, Γκάλ Πέλτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Φέρβερ και για τις δύο εκθέσεις. Τεράστιο το έργο και πολύ καλής ποιότητας. Είναι σαφές πλέον πόσο περίπλοκες και αδιαφανείς έχουν γίνει χρηματιστηριακές δραστηριότητες όπως και τα ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Έχουμε νέα προϊόντα, ε, νέους τόπους διαπραγμάτευσης, ε, νέους τύπους συναλλαγών, αλγοριθμικές συναλλαγές, συναλλαγές ψηλής συχνότητας, έχουν αλλάξει το πρόσωπο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε προς όφελος των πολιτών μας και των επαγγελματιών. Γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο πλαίσιο ενισχύει και εναρμονίζει τις δραστηριότητες ε, των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τις αρμοδιότητες ε, των ρυθμιστικών αρχών με πολύ συγκεκριμένους κανόνες για διασυνοριακή συνεργασία. Είναι σημαντικό οι αρχές ε, να μπορέσουν να ε, καταπολεμήσουν απειλές, κερδοσκοπικές προσπάθειες κλπ. Είμαστε, είμαι υπέρ της ενίσχυσης της ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αγορών και Αξιών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι συναλλαγές ψηλής ε, συχνότητας μπορεί να δημιουργήσουν ιδιαίτερους κινδύνους, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Συνεπώς, πιστεύω θα πρέπει να, έχουμε, να δώσουμε οργανωτικές εγγύσεις ό,τι αφορά τους τόπους διαπραγμάτευσης. Ε, η ε, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση ήταν δυσχερή στο παρελθόν και κάθε φορά που δημιουργούνται αναστατώσει στην αγορά δυσκολεύεται αυτή η πρόσβαση. Πιστεύω ότι οι τόποι διαπραγματεύσεις θα πρέπει ε, να ε, ε, κάνουν ειδικέ εκδόσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να υπηρετούν την οικονομία και όχι το αντίστροφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό η κυρία Μπερέσα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετώντα την έκθεση Φέρμπερ θα μάθει τα πρώτα σημαντικά διδάγματα από την οδηγία MIF 1, υιοθετώντα ένα κείμενο που θα οδηγήσει στην διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενε πλατφόρμε για όλε τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Αυτό λέει αυτό το κείμενο. Το, οι συναλλαγέ ε, υψηλή συχνότητα που μα επιτρέπει σε χιλιοστά το δευτερόλεπτο να εκτελέσουμε μεγάλο αριθμό εντολών θα πλαισιωθεί πλέον από εδώ και στο εξή, γιατί η κρίση έδειξε την ε, καταχρηστική χρήση του, των συναλλαγών υψηλή συχνότητα από κάποιου ε, παράγοντε αγορά που διασάλευαν την λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Η πρόταση του Κοινοβουλίου πάει προς την κατεύθυνση, αποθαρρύνοντα τη χρήση αυτών των πρακτικών και θα ε, βοηθήσει τι χρηματαγορές να λειτουργήσουν ε, προς όφελος της πραγματικής και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Με αυτή την έκθεση το Κοινοβούλιο θέλει επίση να σταματήσει να παρεμποδίσει την κερδοσκοπία στα τρόφιμα που είναι συχνά καταστροφική για πολλού ε, πληθυσμού. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, προσδιορισμοί θέσει και όρια θέσεις για τις συναλλαγές σε πλατφόρμες διαπραγμάτευσης. Η κερδοσκοπία σε πρώτες ύλες ε, γίνεται όλο και πιο πρόδειλη, ειδικά ε, η κερδοσκοπία στα τρόφιμα. Η πρόταση που υιοθετούμε σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα προς σωστή κατεύθυνση στο βαθμό που επιβάλλει όρια στις θέσεις που μπορούν να αναλυφθούν από τους ε, παρεμβαίνοντες στις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης. Αυτή η έκθεση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σημαντικά όταν η Ευρωπαϊκή Αρχή των Χρηματαγορών, ε, Κινητών Αξιών και Αγορών ε, μπορεί να παρεμβαίνει για να απαγορεύσει την πώληση κάποιων ε, χρηματοπιστωτικών προϊόντων που είναι τοξικά και είναι αναγνωρισμένη η καταστατική του συνέπεια στην Ευρώπη. Η σχέση μεταξύ του ΜΙΦ 1 και του κειμένου που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι η εξή. Κατά την εξέταση του ΜΙΦ 1, ε, η βασική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν κυρίως ε, τι θα γίνει με το θέμα των συμβουλών που πρέπει να δίδονται στους ε, επενδυτές και κυρίως στους ιδιώτες επενδυτές, στους μικρούς επενδυτές όταν θέλουν να προβούν σε επενδύσεις. Οι συνθήκε χρηματοδότησης αυτής της συμβουλής είναι ακόμα ένα στοιχείο συζήτησης. Πρέπει να το συζητήσουμε ενδελεχώς ούτως ώστε όλοι ανεξάρτητα από το εισόδημά τους να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ε, συμβουλές μέσα σε συνθήκες διαφάνειας και που θα το επιτρέπουν πραγματικά να κάνει επενδύσεις με τα λόγου γνώσεως όμως. That was too long, too long. Ε, υπερβολικά, υπερβολικά μακροσκελής αυτή η παρέμβαση. Η κυρία Sharon Bowles έχει τώρα το λόγο. Από τους φιλελεύθερους αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της ασφάλεια και του απλώς εντάξει, ασφαλώς θα πρέπει να επιλέγουμε την πιο ασφαλή θέση. Ε, για, τις, τα παράγωγα και την κερδοσκοπία στα τρόφιμα έχουν ακούσει πολλά πράγματα. Ε, εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τις ε, περιορισμένες θέσεις υπό την προϋπόθεση ότι, αν, ότι σε περίπτωση ανάγκης θα μπορούσαν αυτές οι σταθερές λέξεις, οι θέσεις να ε, ε, γίνουν πιο ε, αυστηρές. Έχουμε αυτοματοποιήσει ε, την χαρτογράφηση ε, των ε, συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και αυτό μας βοηθάει να αντιδρούμε γρήγορα. Μας επιτρέπει να παρακολουθούμε κρίσιμες περιοχές όπως η κερδοσκοπία στα τρόφιμα. Και λυπάμαι πολύ που δεν προχωρήσαμε λίγο πιο μακριά σε αυτήν την έκθεση. Έχουμε κάνει καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγαλύτερη δουλειά και σε σχέση με τι ε, ε, προμήθειε. Ε, οι πολίτε θα έπρεπε να είναι σίγουροι ότι παίρνουν τι καλύτερε συμβολέ, όχι ότι σπρώχνονται προ μια κατεύθυνση προ όφελο αυτού που του δίνει τι συμβολές του Συμβούλου. Νομίζω ότι η απαγόρευση θα πρέπει να είναι η, σωστή, η πιο κατάλληλη λύση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόσα Βάγνερ. 1,5 λεπτό. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον ε, εισηγητή και τους άλλους συναδέλφους που συνεργάστηκαν. Η χρηματοπιστωτική κρίση ε, χειροτέρευσε εξαιτία ε, του περίπλοκου συστήματος που συνδέονται με ε, παράγωγα μέσα και εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές με στόχο να αυξηθεί η κερδοφορία πολύ γρήγορα. Ε, ε, μια, ε, είναι πολύ λογικό οι χρηματοπιστωτικές ε, να, κατευθυνθούν προς διαφανείς, διαφανείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης. Είναι απαραίτητο επίσης οι πληροφορίες που δίνονται να είναι κατανοητές από τους επενδυτές που θα πρέπει να γνωρίζουν πλήρως τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να γνωρίζουν και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Δεν έχει νόημα η διαφάνεια ε, ως ε, έννοια αν ε, η διαμόρφωση των προϊόντων είναι τέτοια που δεν μπορούν να τα κατανοήσουν οι πελάτες. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Μάρκους Φέρμπερ για την εξαιρετική του εργασία. Δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα αλλά τελικά καλά τα κατάφερε. Νομίζω ότι η οδηγία MIFID είναι ένα θεμέλιο για τη ρύθμιση των χρηματαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την αναθεώρηση, την αναδιατύπωση της οδηγίας παίρνει σαφή και ε, στεναρή στάση και έχουμε ε, προχωρήσει πολύ περισσότερο από το Συμβούλιο. Θα βελτιωθούν οι δομές, θα μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος, θα ε, βελτιωθεί και η προστασία των επενδυτών και η ΕΣΜΑ θα δει το ρόλο της να αυξάνεται, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Γενικά ε, είναι ε, πολύ καλύτερη κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την παροχή συμβουλών στους επενδυτές, η Επιτροπή ΕΚΟΝ έχει γνωμοδοτήσει. Υπάρχουν μια σειρά ρυθμίσεις ε, για την παροχή συμβουλών με προμήθεια, με αντιπαροχή, καταποκοπή ή δεν μπορεί κανείς να καταδικάσει συλλήβδιν και κατηγορηματικά ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Γι' αυτό ε, είμαι περισσότερο υπέρ της ε, πρότασης Επιτροπής Οικονομικών που θέλει πληροφόρηση και ενημέρωση και διαφάνεια χωρίς να αποκλείει κανένα μοντέλο. Υπάρχουν ε, πελάτες και πολίτες που δεν είναι ικανοποιημένοι όταν ε, η ε, πληρωμή γίνεται με συγκεκριμένη αμοιβή όπως τα ελεύθερα επαγγέλματα. Τι γίνεται με την ενημέρωση και τι γίνεται και με το μάθημα των οικονομικών στα σχολεία. Αυτό θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο για την προστασία των επενδυτών. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και τώρα για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Μακάρθη. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμπερ και τους σκιώδεις ηγητές που έκαναν ουσιαστικές και καινοτόμες βελτιώσεις στην οδηγία για, τις, για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ε, μέσα σε ένα λεφτά θα ήθελα να εστιάσω σε δύο σημασίας σημασία στοιχεία που είναι σημαντικά όμως ε, για την προστασία των επενδυτών και την υπερβολική κερδοσκοπία ε, στις αγορές βασικών προϊόντων. Σε όλη την Ευρώπη οι καταναλωτές ήταν θύματα παροχής κακών συμβουλών λόγω ε, των στρεβλών κινήτρων που ε, προωθεί προϊόντα εις βάρος των βέλτιστων συμφερόντων των καταναλωτών και ε, επενδυτών η διαφάνεια και η πληροφόρηση δεν λειτουργεί όπως έδειξε ένα γερμανικό Ινστιτούτο ε, και αν πληρώνονται αντιπαροχές για συγκεκριμένα προϊόντα τότε οι συμβουλές ε, δεν, ε, δεν τις θεωρούν καλές συμβουλές οι υποψήφοι επενδυτές. Επομένως η λύση είναι όπως στην Δανία, το Βέλγιο, την Δανία κτλ. να απαγορεύσουμε τις αντιπαροχές. Αυτό όμως επέτρεψε στους συντηρητικούς Βρετανούς βουλευτές να ακυρώσουν την απαγόρευση που είχαν ε, επιβάλει οι εργατικοί. Προσοχή λοιπόν πώς αντιμετωπίζουμε την απαγόρευση. Θα πρέπει να κλείσουμε τα παραθυράκια όπου πληρώσαμε άπειρα λεφτά σε έναν ε, ε, κερδοσκόπο ε, στο ο οποίο ε, θα μπορούσε με αυτά τα λεφτά, θα μπορούσε μάλλον με αυτά τα λεφτά να είχαμε θρέψει όλο τον πληθυσμό από το κέρα τη Αφρική κτλ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουλάχ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επαναλάβω εν συντομία ότι το Κοινοβούλιο κάνει καλά τη δουλειά του με την Κομισιόν. Ελπίζω και το Συμβούλιο να κάνει το ίδιο. Είναι, το θέμα είναι ακαθόδε. δύσκολο. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συνεργάστηκε καλά με του Κιώδη. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη δημαγωγία. Μερικέ ε, φορέ μα ρωτούν τι κάνετε για να ρυθμίσετε καλύτερα τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Ε, υποτιμούν αυτά που κάνουμε δεν θα πρέπει να ε, δώσουμε την εντύπωση ότι έχουμε μια μαγική ράβδο που μπορούμε να ε, αλλάξουμε την κατάσταση από την μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην καλύτερη οργάνωση και στην διαφάνεια ε, θα πρέπει σίγουρα να προσπιστούμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Εδώ έχουμε κάποιε μικρέ διαφορέ ανάμεσα στι ομάδε, αλλά γενικά συμφωνούμε. Οι καταναλωτέ θα πρέπει να προστατεύονται περισσότερο. Να προστατεύσουμε επίση και την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Είναι περίπλοκα τα θέματα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί αυτών. Ε, νομίζω, κύριε Επίτροπε, ότι είναι μεγάλη μπουκιά που έχουμε στο στόμα μας. Ε, Χαίρομαι που οι εποπτικές ε, αρχές ε, θα μας ε, βοηθήσουν γιατί και σε αυτόν τον τομέα έχουν πιο αυξημένες μάλλον αρμοδιότητες. Ευχαριστώ κύριο Στόμας Μάν, δύο λεπτά. Η οδηγία MIFID 2, κύριε πίτρο Μπαρνιέ, είναι πραγματικά ορόσημο στο δρόμο προς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των χρηματαγορών. Όλοι οι φορεί θα πρέπει να τηρούν του κανόνε Για να γίνει αυτό χρειάζεται αποτελεσματική, εξασφαλισμένη εποπτεία. Εξού και η εξαιρετική έκθεση του συναδέλφου Φέρμπερ ζητάει προστασία των επενδυτών. Δεν θα πρέπει οι πελάτες μετά από λάθος παροχή συμβουλών να μπαίνουν σε μεγάλο κίνδυνο. Θα πρέπει να δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες και να επιλέγουν εκείνη ε, τη στρατηγική που θέλουν. Και προϊόντα υψηλού κινδύνου θα πρέπει ευθύ εξ αρχής να αναγνωρίζουν και οι αλγοριθμικές συναλλαγές θα πρέπει να ρυθμίζονται καλύτερα και πιο αυστηρά. Τέτοιε συναλλαγές να γίνονται με ταχύτητα φωτός. Ε, αυτό ε, θα πρέπει να σταματήσει. 500 ε, χιλιοστά του ε, δευτερολέπτου θα πρέπει να είναι το ελάχιστο όριο για να μπορούν να ελέγχονται κάπως αυτές οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας. Και αν αυτό γίνεται μόνο για να αυξάνονται τα κέρδη των ε, φορέων, να κληθούν να βάλουν και το χέρι στην τσέπη οι συναλλασσόμενοι. Και χαίρομαι για τα όρια των θέσεων, δηλαδή ε, να υπάρχουν ε, όρια στις συμβάσεις για να μην γίνεται αυτή η υπερβολική κερδοσκοπία με τις πρώτες ύλε. Χρειαζόμαστε τις πρώτες ύλε γιατί είναι ε, μέσα παραγωγής για τη βιομηχανία. Αυτό που σίγουρα δεν χρειαζόμαστε ε, είναι στοιχήματα για τα εμπορεύματα και για την παραγωγή τροφίμων. Και εδώ θα πρέπει να τερματιστεί αυτό με σαφή όρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2009 η ομάδα μου τόνισε τη σημασία των πιο αυστηρών ρυθμίσεων για τις χρηματαγορές. Αυτός ο συμβασμός που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντικό βήμα για μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στη διαπραγμάτευση ψυχολογικής συχνότητας και στην κατάργηση της κερδοσκοπίας στα τρόφιμα. Οι κερδοσκοπικές ε, πράξεις οδήγησαν σε ηλικιώδη αύξηση των τιμών στο παρελθόν για τα τρόφιμα. Ο ο ΦΑΟ, οργανισμός του ΟΗΕ, τόνισε τις καταστρεπτικές συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς στη, και στην, στα τρόφιμα και στο πόσο συνεισέφεραν στην αστάθεια των τιμών των τροφίμων. Η διαπραγμάτευση υψηλή συχνότητα δυστυχώ είναι πάρα πολύ κοινό φαινόμενο στις χρηματαγορές και έκανε μεγάλη ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Υποστηρίζω την έκθεση που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια στι αγορέ. Ο κύριο Λάγκεν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σπάνια έχω την ευκαιρία στην Ολομέλεια να μπορώ να επενώ τόσο πιστικά τον συνάδελφο Φέρμπερ. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ο άνθρωπος. Και ο συμβιβασμό του εγκρίθηκε ομόφωνα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλών διαπραγματεύσεων και πολλαπλών. Πραγματικά θερμά συγχαρητήρια και επένους αξίζει. Θέλω να πω τα εξή τρία εγώ. Πρώτον, αυτό το θέμα με το όριο των θέσεων, position limits. Η λύση που επελέγει, που από ό,τι φαίνεται εφίσταται έξωθεν επιθέσεις, είναι ο σωστός δρόμος. Για να μην καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά γιατί βλέπουμε εκτροπές στα ε, γεωργικά προϊόντα και υπάρχει πρόβλημα με την πείνα στον κόσμο. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες ε, συναλλαγές. Δεύτερον, για το συμβιβασμό που ε, κατατέθη τελευταία στιγμή, για την απαγόρευση των προμηθειών. Έτσι όπως έχει διατυπ μπορεί να αλλάξει σημαντικά την αγορά. Και επειδή εγώ είμαι εισηγητή για τη διαμεσολάβηση στι ασφαλιστικές εταιρείε, θα προτιμούσα αυτό να αφαιθεί στα χέρια των κρατών μελών γιατί υπάρχουν διαφορετικά συστήματα από χώρα σε χώρα. Και να λέμε ότι πρέπει να φροντίσουμε γενικά οι προμήθειε να απαγορευτούν, νομίζω το παρατραβάει. Γιατί ε, αυτό θα σημαίνει κάθε τη συγκέντρωση. Και τρίτον, οι αλγοριθμικές συναλλαγές ή το λεγόμενο εμπόριο υψηλών συχνοτήτων. Και πάλι υπάρχουν πολλοί εδώ από τον κλάδο που είναι κατά του συμβιβασμού. Εγώ συμφωνώ να μειωθεί η συχνότητα των συναλλαγών γιατί στο μέλλον συστήματα υπολογιστών θα χειραγωγούν ακόμα περισσότερο τις χρηματαγορές από ό,τι γίνεται σήμερα. Χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά εδώ. Δεν μπόρεσε αυτό να λυθεί από το MIFID, αλλά στις διαπραγματεύσεις που επίκυνται θα μπορέσει, είμαι βέβαιος, ο εισηγητής να προχωρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δύο λεπτά. Α, όχι, υπάρχει γαλάζια κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε. Ο κύριος Γκίγκολτ. Η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Λάγκεν. Δέχεστε ερώτηση. Okay, fine. Please, the floor is yours. Ε, ε. Κύριε Λάγκεν, εσείς γνωρίζετε ότι ο συμβιβασμός όπως έχει αυτή τη στιγμή δυστυχώς και με θλίβει βαθύτατα δεν φέρνει μεγάλες αλλαγές στο μεγαλύτερο τμήμα των συμβουλών με προμήθεια γιατί οι απαιτήσει διαφάνεια είναι ουσιαστικά ίδιε με τη MIFID 1. Το θέμα είναι η ανεξάρτητη παροχή συμβουλών για τα χρηματοπιστωτικά που στη Γερμανία σχεδόν είναι ανύπαρκτη. Μόνο εκεί ζητείται απαγόρευση προμήθεια. Στα υπόλοιπα παραμένουν όπω ε. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό οδήγησε σε λάθο επενδύσει. Είναι γνωστό ότι ε, μάλλον εσείς ε, το ξέρετε ότι άδικα επικρίνετε τον κύριο Φέρμπερ. Ποιο κύριο Φέρμπερ, δεν τον επέκρινα εγώ τον κύριο Φέρμπερ. Είναι μια συμβαστική τροπολογία που από ό,τι φαίνεται δεν βοήθησαν οι πράσινοι γιατί εδώ ζητάτε ε, υπερβολικά πράγματα. Θα μπορούσε κανείς να γράψει μπορούν τα κράτη-μέλη να φροντίσουν ε, η παροχή συμβουλών επί να Απαγορευθεί; Εγώ θα ήθελα να το αφήσω αυτό στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Και όχι όπως λέει εδώ. Να φροντίσουν τα κράτη-μέλη να απαγορευτεί. Τελεία και παύλα. Να το κοιτάξουν. Δεν καταλαβαίνω οι πράσινοι γιατί δεν το ακολουθούν αυτό. Καθόλου δεν επικρίνω τον κύριο Φέρμπερ. Τους πρασίνους επικρίνω που ζητάνε λαγούς με πετραχίλια. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής. Winkler, δύο λεπτά. Winkler, μάλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Γνωρίζουμε ότι οι μετοχές ε, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση σε κλάσματα του δευτερολέπτου που ε, την αξία τους που τελικά χάνεται. Αυτά δεν είναι ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, είναι καθημερινή πραγματικότητα και έχει τεράστιες επιπτώσεις αυτό στην πραγματική οικονομία και στις εθνικές οικονομίες των κρατών. Και αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι ας το προσπαθήσουμε. Και πολλοί διερωτώνται τι είναι αυτό που ε, ε, μπορεί να σταματήσει αυτή την κερδοσκοπία. Αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να ελέγχεται όσο γίνεται, όσο περνάει από το χέρι μας και αυτός θα είναι ένας από τους λόγους για την αναθεώρηση της οδηγίας. Ε, ε, λύσεις που προτείνονται με τα επιπλέον τέλη, με τους ελέγχους, με διάφορες έκτακτες ρυθμίσεις ε, και μέχρι και διακοπή των συναλλαγών σε όλη την Ένωση. Έτσι θα μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε τους κινδύνους για τις εθνικές οικονομίες. Ε, τι γίνεται με τον καταναλωτή, ε, τι όφελος έχει. Η οδηγία δεν θα πρέπει να ελέγχει μόνο τις αλγοριθμικές συναλλαγές, αλλά να προστατεύει και τους μικροεπενδυτές. Ποιο δεν έχει την αίσθηση ότι ε, εκείνο που τον συμβουλεύει τι προϊόν να αγοράσει τον καθοδηγεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που είναι προ όφελο του πολιτή τελικά και όχι του πελάτη. Χρειάζεται εκεί πέρα μεγαλύτερη διαφάνεια, να ε, υπάρχει επαρκής και διαφανής ενημέρωση για τη συμβουλή και ε, αν είναι αφιλοκερδής, ατελής ή αν υπάρχει προμήθεια θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τα προϊόντα οι καταναλωτέ ανεξάρτητα από την προμήθεια και την αντιπαροχή. Και όλα τα προϊόντα παλιά και νέα να ελέγχονται είναι προς ε, το συμφέρον και το όφελο των πελατών. Και έρχομαι ακριβώ στις προμήθειε να επιτρέπονται μόνο όταν τα γνωρίζει αυτά ο πελάτης όταν είναι απαραίτητες ε, οι προμήθειες για να δημιουργηθεί καν το προϊόν και μετά να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη αν απαγορευτούν συλλήβδη οι προμήθειες και όχι εμεί να το ρυθμίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κύκλο των ομιλητών. Ανοίγει η διαδικασία Catch the Eye. Υπάρχουν δύο συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Δίνω το λόγο στην ε, συνάδελφο κυρία Έλενα Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε τις αδυναμίες ε, στη λειτουργία των χρηματαγορών Υπάρχει σαφής ανάγκη να ενισχύσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα ήθελα να τονίσω ότι ένα παγκόσμιο πλαίσιο είναι απαραίτητο για να εγγυηθεί μεγαλύτερη ποιότητα στις συναλλαγές μας και μεγαλύτερη διαφάνεια. Το εύρος των υπηρεσιών και των μέσων έχει ε, διευρυνθεί τόσο πολύ και όλο και περισσότεροι επενδυτές εμπλέκονται ε, σε αυτές τις αγορές. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει αποτελεσματικό. Οι συναλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε ρυθμιζόμενους τόπους και ρυθμιζόμενες αγορές. Και οι αγορές θα πρέπει να είναι εντελώς διαφανείς. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να καλύπτονται επίσης. Καλώς το βήμα τη συνάδελφο κυρία Ζούμπερ. Τα ευρωπαϊκά όργανα εξακολουθούν να μιλούν για ε, τμήματα της, ε, της ρύθμισης της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Ε, πλην όμως ε, δεν ξέρω αν ε, έτσι καλύπτουμε τις προσδοκίες τις οποίες δημιούργησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν το 2008 παραδέχθηκε ε, ότι, θα, ότι θα λήξουν ε, οι, τα παράγωγα προϊόντα. Προφανώς όχι. Ε, δεν καταπολεμούμε έτσι την κερδοσκοπία. Δεν είναι δυνατόν με τέτοιο αποσπασματικό τρόπο να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία. Το όλο σύστημα βασίζεται στην κερδοσκοπία. Θα πρέπει να αλλάξουμε την ουσία, όχι μόνο ε, την εξωτερική μορφή. Θα πρέπει να καταργήσουμε τα παράγωγα και τους φορολογικούς παραδείσους και θα πρέπει το, η πολιτική εξουσία να ελέγχει την οικονομική εξουσία, να έχει εξουσία επί αυτής. Γιατί αλλιώς τα μέτρα μας θα, είναι ένας ε, κόκκος άμμου σε ένα μηχανισμό ολόκληρο. Ο Επίτροπος έχει τώρα το λόγο. Ο Επίτροπος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα έρθω σε λίγο στην παρατήρηση της κυρία Ζούμπερ. Κυρία Ζούμπερ, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν δίνουμε μερικές απαντήσεις. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Κυρία Ζούμπερ, ασχολούμαστε με κάθε προϊόν, με κάθε τομέα, με κάθε χρηματοπιστωτικό φορέα και παράγοντα όσα χρόνια έχω την τιμή να είμαι επίτροπος, συνεργάζομαι με όλους εσάς και αρκεί να κοιτάξετε τα πράγματα αντικειμενικά. Έχουμε 28 κείμενα κανονιστικά. Αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, ε, όπως φαίνονται σε αυτόν τον πίνακα και εξηγήσετε τα πράγματα στους πολίτες, έχετε την απόδειξη ότι ασχολούμαστε με, όλα τα, με όλους τους τομείς, διδασκόμαστε από τη χρηματοπιστωτική κρίση, κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς οι Ευρωβουλευτές, πέστε το στους πολίτες, έχετε λόγο να είσαστε περήφανοι για τη δουλειά που έγινε από το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προτάσεις αυτές για να διδαχθούμε πραγματικά από την κρίση και να βελτιωθούμε και να κάνουμε αυτό που, που περιμένουν οι πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε τις χρηματαγορές που περιμένουμε όπω είπατε κυρία Γκουλάρ. Σωστά και να είναι αυτέ στην υπηρεσία τη ε, πραγματική οικονομία και όχι να αυτοεξυπηρετούνται όπω τι αφήσαμε να κάνουν περίπου ό,τι θέλανε επί 20 χρόνια. Γιατί το λέω αυτό. Αυτό δεν είναι ένα μου, όπω είπατε. Η έκθεση του κυρίου Φέρμπερ δεν είναι κόκοσά μου. Προτείνει διάφορα πράγματα σημαντικά. Κύριε Κράμερ, ε, κύριε Γκουλάχ, μιλήσατε για την πραγματική οικονομία η πρότασή σας, καθώς και δική μου, ε, δίνει μεγάλη σημασία στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταρχάς, θέλει να δημιουργήσει διαφανείς υγιείς ε, χρηματαγορές, αποτελεσματικές για τη χρηματοδότηση της ε, πραγματικής οικονομίας, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτό που έλεγε ο κ. Στόλογιαν, αυτά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στη χώρα του. Γιατί χρειαζόμαστε πραγματική αξιοπιστία, διαφάνεια, προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών. Επίσης, ε, παίρνουμε και ειδικά μέτρα για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγορές χρηματοδότησης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η ευρωπαϊκή οικονομία χρηματοδοτείται κατά 75% από τις ε, τράπεζες, 25% από τις χρηματαγορές. Είναι μια αντίθετη αναλογία από ό,τι ισχύει στις Ηνωμένες όπου οι χρηματαγορές ε, χρηματοδοτούν 75% της οικονομίας. 25% όμως στην Ευρώπη. Είναι κάτω είναι λιγότερο από αυτό που θα ήθελαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θέλουμε να συνεχίσουμε να, να δουλεύουμε πάνω σε συγκεκριμένα μέτρα για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ε, χρηματαγορές. Με πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις και απαλλαγές, ειδικά για τις βιομηχανικές επενδύσεις. Αυτό το κάναμε με τον κύριο Βέρνερ Λάγκεν στο ΕΜΙΡ και το κάνουμε επίσης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, με τον κύριο με την ε, ρύθμιση για τις τράπεζες. Κύριε Γκέμπελς, ε, μιλήσατε για αυτή τη ρήτρα αναθεώρησης. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι στα περισσότερα κείμενα που, παρα... που παρουσιάζω υποστηρίζω αυτή την ιδέα της ρήτρας αναθεώρησης. Γιατί όπως είπατε και εσείς κύριε Γκέμπελς, αλλά και ο κύριος κύριε κύριε κυρία Μπασέσκου, ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε χρηματαγορές πολύ αποτελεσματικέ πολύ εφάνταστες που χρησιμοποιούν όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά συχνά και τα παραθυράκια, τις τρύπε στην παγκόσμια νομοθεσία και στο παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο. που Πάνε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κινούμαστε εμεί, από τη δημοκρατία κτλ. Και θα πρέπει, όπω είπε και ο κύριο Γκέρβη, να έχουμε αυτέ τι ρήτρε ε, ραντεβού για να επαληθεύουμε και να βελτιώνουμε τα κείμενά μα. Να πω δύο λόγια τώρα για ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό Ξέρετε πολύ καλά ότι ήμουν υπουργό στη χώρα μου για τη Γεωργία και θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Σουίντερν, σε αυτό που υπενθύμησε η κυρία Σουίντερν, Την όλα και μεγαλύτερη α, συμμετοχή των γεωργικών προϊόντων ε, στις χρηματαγορές. Ε, αυτή η συμμετοχή των γεωργικών προϊόντων ε, αυξήθηκε εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Η αστάθεια των τιμών ε, έγινε απίστευτη και με αυτή την, τις ασταθείς τιμές έχουμε πολύ περισσότερα ρίσκα κερδοσκοπία. Κύριε Όλε Σμιτ, κύριε Μακάρθη, κύριε Κλούτον, κύριε Γκέμπελ, κύριε Λάγκεν, κύριε Μπέρε, ο κύριος Τόμα Μάν και κύριος Κούτας, θέλω να σας πω ότι υποστηρίζω τις προτάσεις που έγιναν από τον εισηγητή σα. Ε, για να ενισχύσουμε, κυρία Γκίγκολτ, το, το λέω και σε εσάς, να ενισχύσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Οι προτάσεις της Κομισιόν πάντα ε, επιδέχονται βελτίωσης. Εγώ δεν έχω τη θεϊκή σοφία. Ορισμένα λόγια μου λένε ότι είμαι υπερβολικά φιλόδοξος, αλλά δεν ξέρω τα πάντα. Επιδέχονται βελτιώσεις τα κείμενά μου. Ε, και ευτυχώς το Κοινοβούλιο τα βελτιώνει. Υπάρχει αυτό το θέμα των ορίων θέση, όπου βλέπουμε ότι η διαπραγμάτευση υψηλή συχνότητα πρέπει να πλαισιωθεί. Σωστά. Εγώ δεν θέλω να κάνω πρόταση για να την απαγορεύσω αυτή τη διαπραγμάτευση. Ε, κύριε Γκέμπελ, υπάρχει μια κάποια χρησιμότητά τη για την διαμόρφωση των τιμών, αλλά θα πρέπει να πλαισιωθεί, θα πρέπει να υπάρχουν, υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, να αποφύγουμε τι καταχρήσει. Και ακριβώ αυτό επιδιώκουμε όλοι μαζί. Ε, εξετάζω τι έγινε το Μάιο του 2010 στο flash crash στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, δεν έχουμε καταλάβει δύο χρόνια μετά τι ακριβώς συνέβη τότε. Χρειαζόμαστε αυτήν την αρχή της ευθύνη. Και βλέπουμε, θα δούμε με τη ρήτρα αναθεώρησης αν αρκούν αυτά που προτείνουμε. Ε, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΚΟΝ και η Πρόεδρος Μπόλς τα παρατηρεί όλα αυτά τα φαινόμενα όμως. Ε, μιλάτε για την πλαισίωση των ορίων θέσης πολύ αυστηρή πλαισίωση και θα ήθελα και όλοι οι άλλοι εταίροι του G20, κυρίω οι Αμερικανοί, να επιβεβαιώσουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν το ίδιο. Όλα αυτά ε, με καθησυχάζουν. Η Διεθνής Επιτροπή των Αριθμιστικών Αρχών των Αγορών ε, είπε σε μία έκθεση ότι θα πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω σε αρκετούς ευρωβουλευτές, τον κύριο Όλισμίτ, τον κύριο Μπάλσα, στον κύριο Βάκνερ, Γκίγκολτ, Σουίνμπερν και κυρία Μπερέ για το θέμα των αντιπαροχών, προμηθειών και αντιπαροχών. Ψάξτε να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Πρέπει να ρυθμίσουμε το, τις αντιπαροχές και να τις απαγορεύσουμε εκεί όπου πρέπει να τις απαγορεύσουμε. Προβλέψαμε μάλιστα αυτή την απαγόρευση σε δύο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τις ανεξάρτητες συμβουλές και την διαχείριση χαρτοφυλακίου. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, το να πληρώνεται ο σύμβουλος των προϊόντων είναι απαράδεκτο με τη δυνατότητα παροχής ανεξάρτητης συμβουλής, κάτι που ζητάει ο επενδυτής όμως. Είμαι, έχω απόλυτη επίγνωση τι αλλαγές, σε τι αλλαγές μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια απαγόρευση σε ορισμένε αγορέ και ακριβώς γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν κρατάει τη δυνατότητα οι επενδυτέ να έχουν προσφυγή σε μη ανεξάρτητη παροχή συμβουλών, αν το επιθυμούν. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι σε ένα άλλο κείμενο, στο TRIPS, παράλληλα ε, ενισχύσαμε και απλουστεύσαμε την α, πληροφόρηση που δίδεται και που έχει δικαίωμα να λάβει ο κάθε επενδυτής, ο κάθε ιδιώτης πελάτης. Κύριε Χέλμερ, μίλησατε για τη σημασία του city. Μαζί με το City, το γεγονός ότι έχουμε το City είναι τύχη όχι μόνο για τον Βασίλειο, αλλά για όλη την Ευρώπη. Και δεν καταλαβαίνω, κύριε Χέλμερ, το γεγονό ότι ενισχύουμε την διαφάνεια και ότι προωθούμε ε, υγιεί αγορέ, όπω η οδηγία MIFID επιδιώκει να κάνει, πώ μπορείτε να το θεωρήσετε ω επίθεση στο Λονδίνο. Ήδη καταλαβαίνω πια τι μου γίνεται. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι η υπεύθυνη του City και του Βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν την προσπάθεια που κάνουμε εμείς ε, για την ενιαία αγορά και τι χρηματαγορέ, για τη διαφάνεια και για την πρόθεση υγιών αγορών. Και αν έχω κάτι παρεξηγήσει, διορθώστε με. Κύριε Χέλμερ, είστε υπέρ του φιλελευθερισμού. Θέλω να σα υπενθυμίσω κάτι που θυμάμαι τώρα, απ' δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά. Αυτό που, ο Άνταμ Σμιθ, που ήταν ο πατέρα του φιλελευθερισμού, έλεγε «Δεν υπάρχει αγορά χωρί κανόνε και δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ηθική ε, για, οι φορείς της αγοράς αυτής δεν έχουν ηθική από μόνοι τους. Ε, αυτό προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε ε, αφομοιώνοντας τα διδάγματα της κρίσης. Κύριε Μάρτιν, είμαστε σε φάση συλλογισμού. Μαθαίνουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε μετά την κρίση. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τη θέληση των πολιτών που δεν θέλουν πια να πληρώνουν το κόστος της ρυθμιστικής διαμεσολάβησης και κάποιων ανεύθυνων συμπεριφορών. Συνολικά, κύριε Ευρωβουλευτέ, έχουμε ανάγκη τις χρηματαγορές. Το ξαναλέω μετά την κυρία Γκουλάρ. Χρειάζομαστε όμως ασφαλείς, διαφανείς αγορές και όπως είπε και ο κύριος εισηγητής, μπορούμε να δούμε αν μήπως στις λεπτομέρειες κάτι μας ξέφυγε, αν έχουμε κλείσει όλα τα παραθυράκια, αν έχουμε κλείσει όλες τις ρογμές, ώστε να αφήσουμε όσο δυνατόν λιγότερο περιθώριο στη ρυθμιστική διαμεσολάβηση και να αφήσουμε τη διαφάνεια να παίξει το ρόλο της, αλλά και την ιχνηλασιμότητα. Αυτός είναι ο στόχος που θέλαμε μαζί με τον κύριο Λάγκεν ε, για το κείμενο ΕΜΙΡ. Κυρία Μακάρθη, να σε ευχαριστήσω για τη δουλειά σας, για την έκθεση που μόλις ψηφίσατε για την οδηγία μας που είναι τμήμα αυτού του πακέτου για τις κυρώσεις και τις κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα σε περίπτωση κατάχρησης στις αγορές. Επομένω, είμαστε στην υπηρεσία τη πραγματική αγορά. Θέλουμε οι χρηματαγορές να εξυπηρετούν την πραγματική αγορά και σε όλα τα κείμενα που προωθούμε, σήμερα το MIFID. Το solvency, η φερεγγιότητα, τα συνταξιδοτικά ταμεία μας απασχολεί η πραγματική οικονομία και οι μακροχρόνιες επενδύσεις. Μέσω μιας πράσινης βίβλου θα ξεκινήσει μια συζήτηση. Όχι μόνο πώς θα τιμωρήσουμε τους μακροχρόνιους επενδυτές και την πραγματική οικονομία, αλλά πώς θα τους ενθαρρύνουμε. Και θέλω να στηρίξω τα λόγια που είπε ο κύριος Μπάλτς για την οικονομική διαπαιδαγώγηση των πολιτών. Πολύ σημαντικό, θα το προωθήσουμε με διάφορους τρόπους. Θέλω να συνενώσω και τη δική μου φωνή σε αυτό το χορό συγχαρητηρίων προς τον κύριο Φέρμπερ. Είναι ένα σακρογωνιαίος λήθος σε αυτή την προσπάθεια. Είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο κατοστάρι της επόμενης εβδομάδα. Ευχαριστώ σε όλους. Uh, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής, συνάδελφος κύριος Μάρκος Φέρμπερ. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στα ελληνικά, λέει και Σφέρβερ, αφού ο Πρόεδρος του δίνει το λόγο στα γερμανικά. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομο. Χαίρομαι καταρχάς που έχω τέτοια μεγάλη υποστήριξη από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Δεν ξέρω αν είναι και θετικό αυτό. Καλό ε, είναι που στη μέση βρέθηκε ένα καλό συμβιβασμό. Δεύτερον, να πω ότι εδώ μιλούμε για μια ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, δηλαδή σε ποιες αγορές γίνονται συναλλαγές. Οι συναλλαγές χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Πάντα αυτές οι συναλλαγές έχουν σχέση με κίνδυνο. Δεν υπάρχει χρηματαγορά ελεύθερη κινδύνου και όποιος δαιμονοποιεί τη χρηματαγορά από μόνη της δεν θα είναι ικανοποιημένος με καμία ρύθμιση. Μα δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μας. Η δική μας πρόθεση ήταν να φροντίσουμε αφενός κάθε συναλλαγή με χρηματοπιστωτικά προϊόντα να λειτουργεί και να λαμβάνει χώρα εντός ενός ρυθμισμένου πλαισίου αφενός και αφετέρου αυτές οι χρηματαγορές να δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία και να μην εξυπηρετούν τον εαυτό τους και μόνο. Γιατί αν μάθαμε κάτι από την εποχή πριν το 2008 είναι ότι κάποια στιγμή αυτονομήθηκαν οι χρηματαγορές και δημιουργούσαν προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία και αυτό το ζήσαμε με μεγάλη ε, οδύνη και πόνο το τελευταίο διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και ε, που συνεισέφεραν στην προσπάθεια αυτή. Τους επόμενους μήνες θα τα ξαναπούμε ε, μαζί με το Συμβούλιο και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Και υπό αυτό το καλό πνεύμα που πριτάνευσε τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τον τελευταίο χρόνο, μπορούμε να πάμε στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πολύ και πάλι στα ελληνικά. Κύριε Φέρμπερ, συνάδελφοι, κυρίσω περιομένη τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του συναδέλφου κυρίου Γκοζές με θέμα Ευρωπαϊκή.